Βεβαίως και όπως γνωρίζετε θα προτείνουμε μεταβατικά μέτρα περιορισμένα. Μόνο δηλαδή για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Η ζήτηση ε, του, της έκθεσης του κυρίου Λάγγεν έληξε εδώ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης η έκθεση του κυρίου Στόλογιαν «Συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων». Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον εισηγητή, τον κύριο Στόλογιαν. Έχετε το λόγο για, τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου, στους κοιόδης εισηγητές, ε, στους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων και στα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου που συνεισέφεραν στη συγκεκριμένη έκθεση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτυχή μας συνεργασία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ε, σε τριμερές επίπεδο, των οποίων ε, ηγήθηκε η κυρία Σάρον Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βανίλς, ε, σύμβουλο και υποστηρικτή μας. Σε επίπεδο Μικτών ε, χρηματοπιστωτικών ομήλων υπάρχουν ε, δυνητικοί κίνδυνοι που οφείλονται στην πολυπλοκότητα, στην ε, σύγκρουση συμφερόντων, στη συγκέντρωση και σε άλλους λεγόμενους κινδύνους χρηματοπιστωτικών ομίλων όταν υπάρχουν αρκετές ε, ε, ε, άδειε για διαφορετικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χρηματοπιστωτική όμιλη ετερογενών δραστηριοτήτων θα πρέπει να την χάνουν επιπλέον συμπληρωματικής εποπτείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βελτιώσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για αυτή τη συμπληρωματική εποπτεία σε δύο στάδια. Καταρχάς, ε, ε, το πρώτο στάδιο για να ε, ε, επιδιορθώσει τα πιο τρέχοντα ζητήματα για να επικαιροποιήσει κάποιες υφιστάμενες οδηγίες και η δεύτερη φάση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το 2012 όπου θα προταθεί μια νέα οδηγία για αυτή τη συμπληρωματική εποπτεία για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων που θα βασίζονται σε μια πιο ουσιαστική συζήτηση επί του θέματος αυτού. Μέσω των κοινών μας προσπαθειών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχει καταλήξει τώρα σε συνένεση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την τρέχουσα νομοθεσία σε αυτή τη ε, φάση. Καταρχάς, θέλουμε να καθορίσουμε και να περιλάβουμε τους ε, χρηματοπιστωτικού ομίλους ετερογικών δραστηριοτήτων στη συμπληρωματική εποπτεία, ε, συμπεριλαμβανομένων και των ε, ε, θεμάτων αυτών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, να υπάρχει δυνατότητα τεστ αντοχής σε επίπεδο κάθε χρηματοπιστωτικού ομίλου και να υπάρχει και ε, γενικές κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες θα εκδίδονται από τις εποπτικές αρχές μέσω μιας κοινή επιτροπής. Επίσης ε, θέλουμε να τροποποιήσουμε την οδηγία Φερεγγιότητα 2 και να βελτιώσουμε τη διαφάνεια την ε, συμπληρωματική εποπτείας. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη ε, το δεύτερο στάδιο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο στην έκθεσή μας υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρηση. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει σε αυτή τη συμπληρωματική εποπτεία ε, των μη ε, ρυθμισμένων οντοτήτων κάποια ε, οχήματα ειδικών καθηκόντων. Να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για χρηματοπιστωτικούς ομίλους τους οποίους ε, ε, κατέχουν ευρύτερου όμιλοι που θα περιλαμβάνουν ε, τις συγκεκριμένες ε, διαδικασίες και να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Να υπάρχουν υποχρεωτικά τεστ αντοχής σε επίπεδο μέλλον είναι η τελευταία μας πρόταση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Τώρα ο Επίτροπος ο κ. Μπαρνιέ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στα όσα είπε η κυρία Σάρον και η κυρία Σουίνμπορν επίση μίλησε για συνεργασία περαδελτική και πώς θα ε, συντονίσουμε τι προσπάθειέ μα ε, περί κανονισμών και ρυθμίσεων. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε υπόψη μας ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός ε, τομέας έχει πολλές διαφορές από αυτόν τον της Αμερικής. Καταρχήν, ο τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη χρηματοδοτεί τα 3 τέταρτα της οικονομίας, ενώ στην Αμερική 1 τέταρτο. Βασιλεία 3, Βασιλεία 2 εφαρμόστηκε σε 8.230 τράπεζες, ενώ στην Αμερική μόνο 20 είναι οι τράπεζες, καμία εικοσοριά. Και έπειτα, Άλλη μια διαφορά, και ο κύριος εισηγητής να τον έφερε, είναι το θέμα των ομίλων. Των εταιρικών ομίλων που είναι μια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα. Και γι' αυτό και χαιρετίζουμε την συμφωνία που επετεύχθη για την πρόταση ΦΙΚΟΝΤ και για να σας ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνεργαστήκατε ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κυρίως εσάς κύριε εισηγητά της και τους κοιόδης εισηγητές, την κυρία Μπό, τον κύριο Σκίνερ, Λάμπερτς και Κλούτε. Από την πλευρά του Συμβουλίου θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τι δύο ε, προεδρίε, τη Βελγική και την Ουγγρική, που επέτρεψαν να ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα. Μιλάμε για ομίλους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών που είναι ιδιαιτερότητα ένα επιχειρηματικό πρότυπο το οποίο λειτουργεί καλά. Όμως η κρίση έδειξε πως και εκεί θα πρέπει να ενισχυθούν κάποιες πτυχές της οδηγίας για τους ομίλους αυτούς. Και γι' αυτό και η πρότασή μας έκανε αυτή η Κομισιόν έκανε μάλλον αυτή την πρόταση τον Αύγουστο. Χάρη στη συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο, η υποπτία των χρηματοπιστωτικών ομίλων θα βελτιωθεί ε, καλύπτοντας έτσι ένα αριθμιστικό κενό, συμπεριλαμβάνοντας ε, τα mixed holding, ε, όπως λέγονται, σε τομεακές οδηγίες και στο ε, στην οδηγία αφαιρεγκαιότητα 2 αυτή τη στιγμή θα υποπτεύονται και θα ελέγχονται πιο αποτελεσματικά και αυτό θα οδηγεί στην ενίσχυση πιστεύω και στη σταθερότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ευχαριστώ κυρίως τον εισηγητή σας κύριο Στόλογιαν για τον αποφασιστικό του ρόλο που επέτρεψε την σημαντική βελτίωση σε πολλά σημεία της οδηγίας η οποία, οποία δεν τα είχαμε αρχικά σκεφτά. Α πούμε, το τεστ αντοχή που ανέφερε πριν από λίγο, την ενίσχυση του ρόλου τη Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Αρχών Υποπτία. Όλε αυτέ οι βελτιώσει συμφωνούν με το πακέτο περί εποπτείας. Η συμφωνία επίσης θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας για τις εταιρείε χαρτοφυλακίου. Να χαιρετήσω επίσης και τη συμφωνία που ευρέθη για τη διαφάνεια της δομής των ομίλων αυτών. Εκτιμώ ιδιαίτερα κυρίε και κύριοι τη σημασία που αποδίδει στο θέμα αυτό το κοινοβούλιο. Κάποιες φορές και εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω τις δυσκολίες του Συμβουλίου όσον αφορά την υποχρέωση επικοινωνίας με την Κομισιόν για τους πίνακες ε, που θα δείξουν ε, πώς αυτή η οδηγία μεταγράφει σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό αποτελεί τμήμα των εργασιών μεταγραφής που κάνουν τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, είμαι ευτυχής για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν θεωρεί πως αυτοί οι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειά μας για την καλύτερη νομοθεσία και σας ευχαριστώ που αυτοί οι πίνακες συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο όπως το προτείνετε και όπως αρχικά είχαμε και εμείς προτείνει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ο κύριος Μποντού θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Thank you. of the Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, έπρεπε να ευθυγραμμίσουμε τις προσδιαγραφές και θα ήθελα εδώ να σας πω ότι δεν μπορεί ε, να υπάρξει μία ισότιμη αντιμετώπιση των μεμονωμένων επονδυτών και των τραπεζών και οι δύο κατηγορίες πρέπει να ε, προστατεύονται αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιομορφίες και χαιρετίζω το πρόγραμμα και ελπίζω ότι θα υιοδετηθεί η τροπολογία μου η οποία ζητά να αναβληθεί ε, το ανώτατο επίπεδο της ε, Ρουμανία, για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σε μία περαιτέρω ημερομηνία. Στους ομιλητές εξ ονόματος των ε, πολιτικών ομάδων, ο κύριος Σκίνερ θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Στόλογιαν και τις υπηρεσίες τους και τον κύριο Βανέσο, ο οποίος αναφέρθηκε πολύ συχνά, διότι αποτελεί πάσπαστο τμήμα των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως όλοι σχεδόν προσπάθησαν να βρουν συνένεση για την νομοθεσία αυτή και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε θα επιτρέψει να έχουμε επιπλέον συμπληρωματική ε, εποπτεία για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στη Φερικιότητα 2 και γι' αυτό ακριβώς και χρειάστηκε να νομοθετήσουμε περαιτέρω. Είχαμε και τα αποτελέσματα τα οποία ε, μας έδωσε και η Επιτροπή Διατηλαντικής Συνεργασίας για το θέμα αυτό. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι συμβαίνει όταν όμιλοι εμπλέκονται σε σε πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα και πολύ επικίνδυνα. Ε, για τις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες και άλλες βασικές υπηρεσίες ε, όπου εμπλέκονται τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες σε θέματα ασφαλίσεων υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια αν δεν υπάρχει κατάλληλη εποπτεία τα διατλαντικά ζητήματα είναι ακόμα ζωντανά και μας απασχολούν ακόμα και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει συζήτηση και για τους χρηματοπιστωτικούς ε, ομίλους αυτούς, ε, για τις μικτές εταιρείε, ε, διότι θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά δεν συζητούνται παρκώς και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια πλευρά του Ατλαντικού είναι αυτή η οποία αμφίσταται στις συζητήσεις. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε. Για τα τεστ αντιστοιχή έχετε δίκιο. Ο ρόλο των αρχών, οι πίνακε αντιστοιχία είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικέ επιτυχίε, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και στη συζήτηση σε τριμερέ επίπεδο. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει επιτυχία για τη συγκεκριμένη νομοθεσία, διότι ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, αλλά και των άλλων αρχών στην Ευρώπη, τις οποίες θα πρέπει ε, να περιμένουμε να υποστηρίξουμε. Τώρα η κυρία θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά από την ομάδα των Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ένα βασικό στοιχείο για την εποπτεία των ομήλων είναι η εξασφάλιση ότι αποφεύγεται η επανάληψη της νομοθεσίας. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει ισότιμο πεδίο από την άποψη των διαφόρων τομεακών επιχειρήσεων με τις οποίες ανταγωνίζονται. Αυτά όλα διέπουν σε διάφορες, διάφορες που έχουν υποβληθεί και επίσης όλοι οι κίνδυνοι θα πρέπει να ενσωματωθούν ενώ εξαλείφονται οι επικαλύψεις ε, στην ε, εποπτεία. Αναφέρθηκε ήδη πως ε, όλα αυτά εδώ συμπεριλαμβάνονται και τελικά όλα τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν πως είναι απαραίτητη αυτή η νομοθεσία γιατί διαφορετικά θα είναι περίπλοκη η ένταξή της σε την υπόλοιπη νομοθεσία. Εν γέννη όμως εγώ επαναλαμβάνω πως οι πίνακε αντιστοιχεί είναι σημαντικοί ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Εποπτείας και στην Διοργανική Συμφωνία νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε και ανατομέα αλλά και αναπερίπτωση εξαιρέσεις για τα όσα συμφωνηθούν. Η συμπερίληψη ομοιόμορφων ε, ε, εντύπων αναφοράς μέσα σε δύο χρόνια από την υιοθέτηση των εφαρμοστικών τεχνικών προδιαγραφών επίσης έχει συμφωνηθεί και θα καταστήσει την εποπτεία ευκολότερη. Όπως αναφέρθηκε, οι δοκιμές αντοχής περιλαμβάνονται αλλά δεν είναι ακόμα υποχρεωτικοί και υποχρεωτικές και το να είναι υποχρεωτική περιλαμβάνεται στην ρήτρα αναθεώρησης. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι κάπως απογοητευμένη γιατί το θέμα του πεδίου εφαρμογής περιλαμβάνεται μόνο στην ρήτρα αναθεώρησης, ιδιαίτερα αν δει κανεί τη σημασία ενό μεγάλου ομίλου, παρά να υπάρχει, αντί να υπάρχει ένα απλό κατόφλι. Στην πράξη κάποια κράτη-μέλη μπορεί αυτά όλα να τα ελέγχουν, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην είμαστε πιο τολμηροί ε, σε αυτή την χρονική στιγμή. Όπως είπαν και άλλοι, είναι καλό το αποτέλεσμα, αλλά η επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να είναι πιο τολμηρή. Και το αναφέραμε αυτό σε, για πολλά θέματα που θα θέλαμε να δούμε ακόμα. Τώρα ο κύριος Γκίγκολτ εκ μέρους της ε, ομάδας των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Yeah. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αγαπητέ κύριε Στόλογαν, κύριε Μπανιέ και εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται η έκθεση αυτή κατά τρόπον ώστε να γίνουν οι διορθώσεις ε, σε μία έκθεση που είχε κακώς διατυπωθεί το 2002 σε μία ασαφή οδηγία σχετικά με τους ομίλους όπου υπήρχαν ορισμένα προβλήματα. Καλό είναι να διορθώσουμε τα σημεία αυτά και η κοινή επιτροπή των τριών εποπτικών αρχών δηλαδή ε, των ασφαλιών των τραπεζών και των ε, χρεογράφων να μπορέσουν ε, να συνεργαστούν για ένα γενικότερο θέμα που ξεπερνά τα χρηματοοικονομικά θέματα των ασφαλιστικών εταιριών αλλά βλέπουμε ότι ο διαχωρισμός των τριών αυτών αρχών δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα και στην κατάσταση των αγορών. Έχουμε προχωρήσει και έτσι καταλήξαμε στην ε, ρήτρα αναθεώρηση, στη review clause και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την σωστή έκθεση από τα θεσμικά όργανα και από εσά κύριε Γκαρνιέ και ότι του χρόνου επιτέλους θα μπορέσουν οι πολίτες να λάβουν μία απάντηση στο too big to fail, too interconnected to fail. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε όλο και πιο μεγάλα ε, ε, όργανα που είναι αδιαφανή. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι διάφορες οντότητες που αναφέρονται ως ε, χρηματοπιστωτικοί όμιλοι είναι διάχυτες σε διάφορες τομείς και είναι πολύ δύσκολο να τις διακρίνουμε μόνο σε μία κατηγορία και σε μόνο ένα τομέα της νομοθεσίας πέρασε η κατάσταση αυτή, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές δυσκολίες και η έκθεση που προτείνουμε εδώ οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πρόκειται για ένα κενό το οποίο γίνεται όλο και προφανές ε, σύν το χρόνο. Οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ε, για τις τράπεζες, τις ε, αγορές, θα πρέπει να συνεργάζονται και αυτή η κοινή μεικτή επιτροπή μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα. Θα πρέπει να υπάρχει ε, πιστοποίηση και παλήθευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της εφαρμογής αυτής της οδηγίας για να μην υπάρχουν ε, πιθανές ε, που θα διακυβεύσουν την ασφάλεια και τις εγγυήσεις στον τομέα. Η αλληλεξάρτηση που δημιουργήθηκε στο χρηματοπιστωτικό τομέα χρειάζεται σαφώς νέους κανόνες οι οποίοι θα είναι πιο έγκαιροι και πιο εκτεταμένοι ε, για να μην καταλήξει να χρεοκοπήσει όλη η ευρωπαϊκή διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ζητήσω να λάβει το λόγο η κυρία Έλενα Μπασέσκου. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω ε, συγχαίροντας το συνάδελφο Στόλο Γιάν διότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία συμπληρωματική εποπτεία για να μειώσουμε τους κινδύνους και οι οντότητες οι οποίες ανήκουν σε ε, ένα όμιλο χαρακτηρίζονται από την παγκοσμιοποίηση που επέδρασε σε όλους τους τομείς και απέδειξε ότι δεν επαρκούσε η εποπτεία στο χρηματοοικονομικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να αποβλέπουμε ε, την ε, ε, παρακολούθηση των μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων που δεν ε, μπορεί ε, κανείς πάντοτε να παρακολουθήσει χωρίς όμως να διαχωρίζουμε τις τραπεζικές από τις ασφαλιστικές εργασίες. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία εναρμονισμένη εποπτεία κατά τρόπον ώστε να ενισχύσουμε και τους σχετικούς οργανισμούς. Θα συνεχίσω ουγγρικά.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 και στο μέλλον θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ηρεμία στις χρηματαγωγές και ως εκ τούτου να αλλάξουμε την ε, οδηγία και να ε, εκπονήσουμε μία νέα οδηγία για την συμπληρωματική εποπτεία κατά τρόπο ώστε να μπορέσουμε ε, να μειώσουμε τις επιπτώσεις των οργανισμών αυτών στη γενική αγορά. Ευχαριστώ την ε, ομιλήτρια και δίνω το λόγο στον Ζων Πολ Γκοζές. Κύριε Πρόεδρε, έχω να κάνω μία παρατήρηση και μία αίτηση. Καταρχήν η παρατήρηση είναι ότι χάρη στην εργασία του κυρίου Στόλογιαν ε, καταλήξαμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση που θα προωθήσει ή στο Συμβούλιο για να ε, δοθεί συνέχεια στους τρεις άλλους τομείς και ε, θέλω να δώσω τον κύριο, ε, το λόγο στον κύριο Μποντούς σαν συντονιστή της ομάδας ε, ΕΛΚ ο οποίος προηγουμένως έκανε μία αναστροφή σχετικά με τα σχόλια που έκανε ονόματι της νομικής επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμπληρωματική εποπτεία θα πρέπει να λάβει και υπόψη και του συστημικούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι στην αγορά. Η συμπληρωματική εποπτεία θα είναι επιπρόσθετη και δεν ε, θα καλύπτει την εποπτεία που θα κάνουν τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις ε, αγορές των τραπεζών και τις ασφαλιστικές αγορές επίσης. Θα πρέπει να γίνεται εποπτεία σε επίπεδο ομίλου. Η συμπληρωματική εποπτεία δεν θα δώσει επιπλέον γραφειοκρατία, διότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών, ώστε να γίνεται κατάλληλος καταμερισμός των αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά. Ο κύριος Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και ο εισηγητής έχει δίκιο ότι πέρα από την καταπολέμηση των συνεπειών της κρίσης, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κατάλληλη νομοθεσία για να διορθώσουμε για την ρίζα του κακού. Αυτό είναι λοιπόν ένα σωστό, μια σωστή προσέγγιση. Καλύτερο έλεγχο των κεφαλαϊκών ροών θα πρέπει να είναι μια από τι πολιτικέ μα. Θα πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. για να δούμε ακριβώς και σε για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά. Ε, θεωρώ ότι έληξε η διαδικασία Catch the Eye και παρακαλώ τον ε, Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, κλείσει τη συζήτηση επί του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές οι οποίοι εκφράστηκαν ε, και ακολούθησαν τη γραμμή του κυρίου Στόλογιαν. Θέλω όμως να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και ορισμένες διευκρινήσεις. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Σκίνερ που είναι ειδικό στον τομέα και εγώ σκέφτομαι κύριε Σκίνερ ότι θα ενισχυθεί κατά αυτόν τον τρόπο η ολοκληρωμένη συμπληρωματική εποπτεία και πιστεύω και εγώ ότι είναι μέρος του προγράμματος του G20 που έχω αναφέρει επανειλημμένως στις συζητήσεις μας και πιστεύω ότι κανένα προϊόν, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν πρέπει να διαφεύγει από μία έξυπνη εποπτεία. Ο κύριος Ικίρσκι τώρα μόλις ανέφερε το θέμα της συνολικής εποπτείας. Ε, κύριε ε, Σκίνερ, σχετικά με τη συζήτηση που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, σας είπα πόσο χρόνο αφιερώνω και προχωρούμε. Το κείμενο το οποίο ανέφερε προηγουμένως ε, ο κύριος Λάνιν για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα απετέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων τεχνικών με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Κύριε Σκίνερ, μπορώ να σας πω ότι η συζητήσεις αυτές είναι έντονες, ε, επικοδομητικές και τίποτα δεν παραβλέπεται. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο και το ανέφερα προηγουμένως σαφώς, ε, το ανέφερα επίσης ή στον Αμερικανό Υπουργό και του είπα ότι το θέμα αυτό που είναι ιδιαίτερο για τους Ευρωπαίους θα καλυφθεί και θα εξαντληθεί από δικής μας πλευράς στην επεξεργασία του. Δεν σημαίνει ότι δεν αναλωνόμαστε στον διατλαντικό οικονομικό διάλογο αλλά ε, μιλάμε εδώ για τη Συμφωνία της Βασιλείας διότι ότι μιλάμε για τους global traders όπου παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις. Όντως το αποτέλεσμα που επιτύχαμε είναι καλό χάρη σε εσά σχετικά με τους πίνακες συσχετισμού και χάρη στη συνεμνία η οποία γίνεται στο κείμενο. Πρέπει να πω στον κύριο Γκίγκολντ ότι όντως πιστεύω ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ε, αντιμετώπιση και αυτό το είπε και ο κύριος Μοργάν είναι ένα θέμα διαφο... Ε, σημαντικό και γι' αυτό όλοι μαζί προβλέψαμε μία αναθεώρηση για το 2012-2013 το ταχύτερο δυνατόν. Κύριε Κίγκολτ, ούτως ή άλλως αυτά τα μέτρα είναι μόνο το πρώτο βήμα. Θα προχωρήσουμε στα πλαίσια των ομίλων και εντός ε, του πλαισίου της εποπτείας ε, σε αυτό το θέμα και ελπίζω ότι σε μερικά χρόνια θα καταλήξουμε σχετικά με με το CRD4 και με το πακέτο Φερενγκιώτης 2. Το πρόγραμμα λοιπόν το οποίο είναι ειδικό για την Ευρώπη και πλήττει όλους τους ισχυρούς θα μπορέσει να ενισχύσει την εποπτεία των ομίλων το 2012 και 2013 και όπως είπε και η κυρία Μπολ θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν τολμηρότεροι. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο Θεοδόρ αν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Για όλα όσα ακούσαμε σε αυτή τη συζήτηση, προέκυψαν κάποια θέματα για τα οποία έγινε μακρά συζήτηση στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Οι συνάδελφοι πρότειναν και κάποια θέματα εν είδη τροπολογιών και το βασικό πρόσκομα το οποίο αντιμετωπίσαμε και δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί των θεμάτων αυτών ήταν το γεγονό ότι δεν υπήρχε αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι συζητάμε το χρηματοπιστωτικό τομέα, ένα τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο για κάθε νομοθεσία και κάθε ε, ε, νομοθέτημα έχει κάποιο κόστος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προτείνουμε νομοθετήματα για ε, οντότητες που προδραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου να είναι σε θέση να προτείνει μια νέα οδηγία για τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομήλων όπως μας έχει υποσχεθεί και θα ήθελα ε, για μια τελευταία φορά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Μπαργινιέ και το προσωπικό του, το οποίο εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και συνεργάστηκε με την Ουγγρική Προεδρία και με τους συναδέλφους μας προκειμένου να καταλήξουμε στη συνένεση η οποία ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Θα Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Tisztelettel közlöm a plénummal, hogy ezennel a vitát berekeztem, και a szavazásra holnap déli...